Karp tego 10 sekund w Kazachstanie trzeba dowiedzieć, dobrze? Please sit down. Dear colleagues, ladies. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε στις θέσεις σας. Αγαπητοί φίλοι, παρακαλώ, το γρηγορότερο δυνατόν να καθίσετε στις θέσεις σας.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 Ε, Αγαπητοί φίλοι, σε ένα λεπτό θα αρχίσω. Καθίστε παρακαλώ. Otwieram posiedzenie. Άρχεται η συνεδρίαση. θα ήθελα να σας υπενθυμίσω